επανάληψη της Συνόδου. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης είναι διαθέσιμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσεις κατά των πρακτικών αυτών. Ενστάσεις. Όχι. Θεωρούνται εγκεκριμένα λοιπόν. Κυρίε και κύριοι, το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη